άλλη χώρα χωρίς να τηρούν τους κανόνες. Χωρίς κανόνες λοιπόν ήταν δυνατόν να αναζητήσει κανείς ε, βραχυπρόθεσμα κέρδος και να εγκασταθεί στη χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς και τους λιγότερους φόρους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κανόνες οι οποίοι θα προστατεύουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Η προστασία στα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβουλεύσεων, η προστασία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στη συνάδελφό μου την κυρία Ρίγνη ε, για την επιτυχία που σημείωσε παρά τις δυσκολίες. Η πρώτη επιτυχία της είναι ότι πλέον από μια χαόδη κατάσταση περνάμε σε μια ρυθμιζόμενη ε, η διοίκηση για πρώτη φορά είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στο προσωπικό ένα, μια λεπτομερή έκθεση ε, σχετικά με την αναδιάρθρωση της εταιρεία. Μια ρήτρα κατά των καταχρήσεων θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν τα αίτια της αναδιάρθρωσης. Καλό και έτσι λοιπόν ε, η ε, εξελίξεις αυτές και τα φαινόμενα των εικονικών εταιριών μπορούν να αποφευθούν. Τα κράτη-μέλη βέβαια δεν ήθελαν να κάνουν άλλο ένα μεγαλύτερο βήμα, έχασαν αυτή την ευκαιρία. Αλλά δεν ήταν η Ευρώπη, δεν ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών που είχαν παρεμποδίσει, που παρεμπόδισαν την καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Το Κοινοβούλιο βρήκε καλές συμβαστικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές δείχνουν το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και στο θέμα της συναπόφασης. Βλέπουμε να υπάρχει μια πλήρης αντίφαση ανάμεσα στα συνδικαλιστικές, ελευθερίες και στα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Το κείμενο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι η καλή αρχή για ένα σύστημα κανόνων. Εγώ θα υπερψηφίσω το κείμενο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι επιγόντως απαραίτητο να υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο για τη συναπόφαση επειδή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωπαίους πολίτε, αλλά και τους συναδέλφου μου για το ότι μου έδωσαν τη δυνατότητα να εργαστώ και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τέτσερ και καλή τύχη. Ο κύριος Σίτερβαν τώρα για την ΚΟΕ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους εισηγητές που αγωνίστηκαν ε, κατά της φοροδιαφυγής ε, και υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά διαπιστώνω ότι ένα πολύ καλό κείμενο του Κοινοβουλίου νοθεύτηκε στον τριμερή διάλογο. Αυτό το οφείλουμε στο Συμβούλιο που δεν είναι παρόν. Υπάρχουν νέοι κανόνες ε, για το δικαίωμα εγκατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους νέους κανόνες δυσχεραίνεται η ε, άσκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ε, εμείς θέλαμε να αποφύγουμε τις εικονικές εταιρείε, ε, να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωτικότητα. Καλό αυτό, όμως ε, χάνονται τα δικαιώματα των πολιτών, γίνεται κοινωνικό ντάμπινγκ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως αριστεροί, όπως και ο συνάδελφος, ζητάμε μια οδηγία πλαίσιο για τη συναπόφαση, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ο κύριος Βόμποντα απουσιάζει, Επομένω το λόγο έχει ο κύριο Ράντεφ. Έχετε ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σήμερα συζητάμε αυτό το νομοθετική πράξη που αποτελεί μέρος του εταιρικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ρέγνερ αλλά και την Κομισιόν γιατί άκουσε την εκκλησία μας για διασυνοριακή εναρμόνιση σε περίπτωση των μετατροπών συγχωνεύσεων και διασπάσεων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο κύριος σκοπός είναι να διευκολύνουμε τις ε, εταιρείε και κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν προβαίνουν σε μετατροπές, ε, συγχωνεύσεις και διασπάσεις διασυνοριακά. Η οδηγία αυτή θα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό. Ο έλεγχος καταλληλότητας, πιστεύω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υποχρεωτικά μέτρα κατά της κατάχρησης θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να σταματήσουν ε, κάποιες τέτοιες πράξεις όταν ε, έχουν ε, απατηλό σκοπό. Εδώ έχουμε διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα των πιστωτών, των μετόχων και των εργαζομένων. Οι εργαζομένοι θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τις συνέπειες των διαδικασιών αυτών και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και όσων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου θα προστατεύονται. Ταυτόχρονα οι πιστωτές θα έχουν ε, ξεκάθαρες ε, και αξιόπιστες εγγύησεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ράντεφ. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών και δεν υπάρχει κάποιος ομιλητής για τη διαδικασία Catch the Επομένως θα δώσω τον Επίτροπο στην κυρία Γιούροβα. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρεμβάσεις σας για τα θετικά σας σχόλια. Ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς όσους τονίσατε ότι χρειάζονται κανόνες για την καλύτερη κινητικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες. Πράγματι αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έχουμε αυτή την νομοθεσία διευκόλυνσης η οποία θα ε, παρέχει και ασφαλιστικές δικλείδες κατά της κατάχρησης, ασφαλιστικές δικλείδες που θα εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων των μετόχων ε, και των εργαζομένων, που θα εγγυώνται ότι δεν ε, θα έχουμε φοροποφυγή, φοροδιαφυγή ή τη δημιουργία εταιριών προπετασμάτων, εταιριών γραμματοκιβωτίου. Ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη αυτή η νομοθεσία, χρειάστηκε πολύ εμπειρογνωμοσύνη και όπως είπα και στην αρχή, χρειάστηκε και μεγάλη πολιτική βούληση. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι συνεργαστήκαμε σε ένα πνεύμα συμβιβασμού. Και βέβαια μας πίζει και ο χρόνος ε, στο τέλος. Είμαστε στο τέλος της θητείας μας, αλλά τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεργασία. Πιστεύω ότι από κοινού παρουσιάζομαι μια καλή και ισορροπημένη πρόταση και ελπίζω ότι αύριο θα υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιούροβα. Η Εβελίν Ρέκνε τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όποιος ε, έχει ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο ε, πρέπει να είναι μαραθωνοδρόμος με ε, ικανότητες ταχείας με ικανότητες πρινταρίσματος όπως τα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο εμείς Ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια για να επιτύχουμε καλές προδιαγραφές στην Ευρώπη. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιότητα και μέχρι και το τέλος, μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας αγωνιστήκαμε για να περάσει η δέσμη μέτρων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο, ε, τους ε, διαπραγματευτές από τη Ρουμανική Προεδρία, την Γκαμπριέλα συγκεκριμένα, να ευχαριστήσω ε, τους ε, σκιώδης ηγητές και κυρίως και τους συνεργάτες μας. Θα ήθελα αυτό το τελευταίο λεπτό να το εκμεταλλευτώ για να πω ότι ναι πράγματι έχουμε τώρα επιτύχει πάρα πολλά και σημαντικά αλλά το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η οδηγία πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα οριζόντιο εργαλείο για τους εργαζόμενους έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε και το περίφημο escalator έτσι ώστε να μπορεί να γίνει, να υπάρξει προσαρμογή ανάλογα με τις ε, καταστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε ε, και σας συζητήτρια και την Επίτροπο έκλεισε η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Και συνεχίζουμε στην εμερήσια διάταξη και φτάνουμε τώρα στην ε, έκθεση του κύριου Στίσλαβ Κρασνοντεύσκη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή πρώτα. Παρακαλώ. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Γιατί μετά από τρεις τριμερείς διαλόγους και ώρες διαπραγματεύσεων, καταφέραμε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια μερική συμφωνία που θα ψηφιστεί αύριο. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Εκφράστηκαν πολλοί φόβοι για το ταμείο αυτό. Φόβοι που εμένα μου φαίνεται ότι δεν έχουν καμία βάση. Αυτοί οι φόβοι, αυτές οι διαφωνίες, οι αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα κάτι το οποίο μένα με εκπλήσει. Εγώ προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, όλων των συναδέρφων του κύριου Μπούτικοφερ, για παράδειγμα, του κύριου Μαρτά, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τα επιχειρήματά τους και είχα την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι αυτοί ήταν λίγο πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θέτουν υποαμφισβήτηση το κείμενο αυτό και βασίζονται ε, στα εξή δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι ηθικής και το άλλο έχει να κάνει με τη φύση της κατεξοδότησης πράξης. Το ζήτημα ήταν, όσον αφορά την ηθική πτυχή, το μήπως το Ταμείο αυτό αμφισβητεί τις σχέσεις μας με την Ατλαντική Συμμαχία, με το ΝΑΤΟ, που αποτελεί και την δομή που μας εγγυάται την ασφάλειά μας. Αυτό ερχόταν μάλλον από το αριστερό τμήμα του ημικυκλίου. Ακόμα και αν υπήρχαν ε, τέτοιες φωνές που ακούστηκαν και από το κέντρο και από τη δεξιά πτέρυγα του ημικυκλίου. Αυτά τα επιχειρήματα δεν έχουν βάση. Ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε πιστεύω ότι αναγκάζει το Συμβούλιο να σέβεται απόλυτα τα όσα διαπραγματευτήκαμε. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι η Επιτροπή, η Επίτροπος, είναι ικανοποιημένη και αυτή από τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Επιτρέψτε μου τώρα να παριθμίσω κάπως γρήγορα τι πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλο ότι το Ταμείο αυτό θα το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, ότι η τεχνολογία θα διακρίνεται, ότι το επιπλέον ο κόστος δεν θα περιορίζεται, ότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις προτιμησιακές στη συμμετοχή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και εκείνες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επίσης ότι θα υπάρχουν απαιτήσει ηθικής πάρα πολύ αυστηρές για οποιαδήποτε δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο αυτό. Συνεπώς, πετύχαμε πολλά από το Συμβούλιο. Αν συγκρίνουμε, δηλαδή, ό,τι προβλέπεται για το Ταμείο από το ΕΔΙΤΠ, αυτό που είναι, ας πούμε, για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πετύχουμε ότι επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος αν υπάρχουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείονται από την χρηματοδότηση. Επίσης πετύχαμε ότι η αναφορά για στήριξη από το Ταμείο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί έτσι δείχνουμε ότι το Ταμείο δεν θέλει να στρατιωτικοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να προωθήσει τις εξαγωγές όπλων. Όχι. Θέλουμε να στηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον ε, τομέα των εξοπλισμών. Και είμαι πεπισμένος ότι το Ταμείο αυτό θα επιτρέψει να δημιουργήσουμε νέα τεχνολογία και άμυνα υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που δεν καταφέραμε όμως να πετύχουμε από την άλλη μεριά εννοείται είναι μέσα στη φύση του Ταμείου, είναι η κατεξιοδότηση πράξη. Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί το Ταμείο από την αρχή του 2021. Ίσως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να αναφέρει κανείς, αλλά εγώ αυτά ήθελα να πω μέχρι τώρα. Διατηρήσαμε τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά επιχειρήματα αυτά της αριστεράς δεν στέκουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ε, ε, εκ μέρους ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο πρόεδρος ο κ. Μακάλιστερ. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο κάνουμε ένα μεγάλο βήμα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα κοινά στοιχεία στην ε, έρευνα και στον, ε, στην αγορά ε, στρατιωτικών εξοπλισμών. Έτσι για να μπορούμε να οργανώσουμε την άμυνά μας. Ως εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό, ένα πράγμα κρίνω ιδιαίτερα σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θέτει τα θεμέλια για καλύτερη συνεργασία και πάνω σε αυτό ε, μπορούμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω σε θέματα ασφάλειας, ε, πολιτικής ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση των ε, εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη στρατιωτική ικανότητα και σε τελική ανάλυση μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους φόρους. Με το αμυντικό ταμείο βελτιώνουμε την αμυντική μας ικανότητα και ως εκ τούτου και την προστασία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν Λοιπόν, καλώ όλους τους συναδέλφου αύριο το μεσημέρι να υπερψηφίσουν αυτόν τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, ε, κύριε Μακάλιστερ. Τώρα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Πιανκόφσκα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, για άλλη μια φορά χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία ή που μας δίνετε ευκαιρία να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο δεν υπάρχει συνεργασία για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Η πρόταση της Επιτροπής, από τότε που υπήρξε αυτή η πρόταση, είχαμε πολύ ουσιαστική δουλειά. Ε, σήμερα έχουμε μία ψηφωνία για την οποία ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αύριο. Τα βασικά στοιχεία του Ταμείου αποτελούν ορόσημο για την Μυντική Ένωση. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να ευχαριστήσω την ε, διαπραγματευτική ομάδα τη ΙΤΡΕ. Όλοι σα ε, είσαστε πολύ αφοσιωμένοι. Ο εισηγητή, η κυρία Γκροστέ, το κύριο Ρικέ, Μαρτάν Μπιουτικόφερ και βεβαίω ε, δεν πρέπει να ξεχνάω και τον κύριο Μακάλιστε. Σα ευχαριστώ όλου σα θερμά. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θα ενισχύσει την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, θα βελτιώσει την αμυντική της ικανότητα και από την άλλη ε, θα βελτιωθεί η χρήση των ε, δημόσιων κονδυλίων. Με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευαισθητοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά και να επιφέρουμε καινοτομίε ε, βελτιώνοντας ε, την τεχνολογική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος κάνοντας την Ευρώπη μια πηγή ασφάλειας, ε, όχι σε αντίφαση με τον ΝΑΤΟ, αλλά συμπληρώνοντάς του. Θα περιλαμβάνονται πάρα πολλά στοιχεία Γι' αυτά αγωνίστηκε σκληρά το Κοινοβούλιο. Θα αναφέρω λίγα εξ αυτών. Τα ανέφερε ο συγητή, αλλά θα τα πω και εγώ από την προοπτική τη Επιτροπή. Πρώτον, οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωσης θα ισχύουν με βάση τον κανονισμό και την ενωσιακή ε, διακυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Ε, το ε, Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτό το Ταμείο. Δεύτερον, θα ε, τεθεί το θέμα της ε, επιλεξιμότητας σε σχέση με το Ταμείο. Εδώ οι κανόνες είναι σαφείς. Μόνο οι ενωσιακές ε, εταιρείε, οι οποίες σέβονται θέματα ασφάλειας στον εφοδιασμό και σε πολλούς άλλους τομείς, μόνο αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανένα, απλά ορίζουμε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή για να διασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλίζονται τα συμμετοχή συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές εταιρείε όταν ασχολούνται με έρευνα και ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. Τρίτο θέμα, συνεργασία. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του Ταμείου. Εμείς δίνουμε κίνητρα με συγκεκριμένους κανόνες, προκαλώντας και την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους αμυντικούς ομίλους, αλλά και μικρούς παίκτες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς ελπίζουμε να ανοίξουμε την αλυσίδα την αμυντική. Τέταρτον, στο νομικό κείμενο καθίσατε σαφές ότι οι πράξεις θα πρέπει να είναι συμβατές ε, με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, όπως επίσης και με ηθικές αρχές που περιλαμβάνουν τα δίκαια αυτά. Το Κοινοβούλιο ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ε, εκφραστεί επί των θεμάτων της δεοντολογίας και επί των εμπειρογνωμόνων. Επίσης, το Ταμείο αποκλεί δράσεις ε, για την ανάπτυξη θανατηφόρων όπλων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Εξάλλου, εμείς θα στηρίξουμε τις καινοτομίες το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό ε, βρίσκονται στην ίδια θέση, κυρίως αφορά τις αποκαλούμενες disruptive ε, τεχνολογίες. Αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Σιγητή ότι ε, θα έχουμε τις εφαρμοστικές πράξεις Έχουμε έναν κατάλογο που εισήχθη για να οριστεί το πλαίσιο του προγράμματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη και πρόθυμη να έρχεται κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο για να συζητιέται το πρόγραμμα. Αυτή η προσέγγιση δεν αφορά μόνο θέματα άμυνας. Υπάρχουν και άλλα ε, προγράμματα και άλλες προτάσεις χρηματοδότησης που καταφεύγουν σε εφαρμοστικές πράξεις και που γίνονται δεκτά από το Κοινοβούλιο και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Μπιενκόφσκα. Στην ε, συνέχεια, από την Επίτροπη Προπολογισμών, ο κύριος Λαμασούρ. Για ένα λεπτό, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι εξ ονόματος Επιτροπής Περιπολογισμών, ε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους ε, όσους πέτυχαν αυτή την μερική συμφωνία και ιδίως την ομάδα του Κοινοβουλίου η κυρία Επιτροπό ανέφερε τα μέλη τη για την Επιτροπή Προπολογισμών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο ενωτόμα ε, έργα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια προκειμένου η άμυνα να μπορεί να αποφεληθεί από κονδύλια της Ένωσης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η συμφωνία αυτή δίνει στο πρόγραμμα όλα τα μέσα για να πετύχει τη φιλοδοξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα μέσα του InvestEU και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αύριο θα το επιβεβαιώσει η Ολομέλη. Επίσης, χαίρομαι για το πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα που στέλνει αυτό το πρόγραμμα σε ένα τομέα που βρίσκεται στην καρδιά της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό το ταμείο μας δείχνει ότι η μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων ταχυτήτων στη συνένωση θα επιτρέπει να έχουμε περισσότερη ασφάλεια για να έχουμε και μικρότερο συνολικό κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμασούρ. Στη συνέχεια, εκ μέρου του ΕΛΚ, η κυρία Γκροστέτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο κύκλο αυτό μετά από 20 ετή παρουσία και είμαι ικανοποιημένη που μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμήνα απόψε, γιατί ελπίζω ότι θα είναι ένα επιπλέον εργαλείο ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω τη ανάπτυξη τη συνεργασία. Πρόκειται για ιστορική στιγμή και αποφαλούμε να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κρασνοντεύσκη και την Επίτροπο, την κυρία Μπιένκοφσκα, που μας επέτρεψαν να πετύχουμε μια ταχεία συμφωνία. Ε, βέβαια, κάποιοι προσπάθησαν να κάποιοι να μπλοκάρουν ε, τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε πραγματική βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμενος και κάτι που κανείς δεν φανταζόταν δυνατό, το πετύχαμε έτσι λοιπόν. Ε, έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία που πρόκειψε από τις διαπραγματεύσεις και ε, στο επόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει τον προπολογισμό των 13 δισεκατομμυρίων την περίοδο 2021-2027. Θα πρέπει να προσελκύσουμε τα καλύτερα προγράμματα και τα πιο καινοτόμα από την πλευρά των κρατών μελών και τη βιομηχανία. Αυτό το ταμείο απαντά στις ανησυχίες των πολιτών μας για την ηθική, για την απαγόρευση των θανατηφόρων οπλικών συστημάτων. Έχουμε επιχειρήματα απέναντι σε κάποιες ειρηνικές ε, ιδεολογίες που ε, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Αυτό το Ταμείο θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ενισχύσει την αυτονομία της σε στρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μία ανεξάρτητη ικανότητα με χρηματοδότηση προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσει. Αυτή η αρχή τη στρατηγική αυτονομία, είναι ζωτική σε πολλού άλλου τομεί, στο διάστημα, στην υγεία, την ενέργεια, τα τρόφιμα και βεβαίω στην ασφάλεια και στην άμυνα. Γιατί σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο θα πρέπει να βασιζόμαστε στην ένωση με τι δικέ μα δυνάμει. Έτσι θα έχουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτρέψει να προστατεύσει καλύτερα την ασφάλεια των κρατών μας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κροστέτ και σας ευχόμαστε ότι καλύτερο στο μέλλον. Είπατε μετά από 25 χρόνια είναι η τελευταία σας παρέμβαση αυτή. Ωραία. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Εντουάρ Μαρτά, παρακαλώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως και καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο κατάφεραν να φτάσουν σε αυτήν την συμφωνία και χαίρονται, αυτό θέλανε και δεν υπάρχει κατεξουσιοδότηση πράξη. Κάτι που μπορεί να φαίνεται ένα τεχνικό στοιχείο για πολλούς, αλλά όχι, γιατί είναι θέμα ελέγχου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα των πολιτών για ένα πρόγραμμα 13 δισεκατομμυρίων και για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Φυσικά και στηρίζω τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε αύριο και ιδιαίτερα το άρθρο για την απαγόρευση κάποιων όπλων, το άρθρο 11 επίση, γιατί πράγματι δεν είναι δυνατόν απλώ να αναφερόμαστε στο διεθνέ δίκαιο, γιατί υπάρχει εμφυσιμία εδώ. Για παράδειγμα, ο λευκός φόσφορο, η χρήση του για πυρομαχικά επιτρέπεται. Αν όμως χρησιμοποιηθεί χωρίς ε, διακρίσεις εμπριστικά, αυτό το καταδικάζει η ίδια σύμβαση της Γενέβης. Και έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις που έχει καταδικάσει ε, ε στην Γάζα, για παράδειγμα. Έπειτα, το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Και εδώ, σαν όπλο, απαγορεύεται στο Βέλγιο. Δεν ρυθμίζεται όμως αλλού και ούτε αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο. Εφόσον λοιπόν ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται, θα έπρεπε να έχουμε ένα κατάλογο με συγκεκριμένο εξοπλισμό για τον οποίο δεν πρέπει να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, για τι εξαγωγέ όπλων. Δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυρώνει την προσέγγιση που θέλει το Συμβούλιο να είναι όλα στην διακριτική ευχέρεια των χωρών μελών. Είναι θέμα ερμηνεία. Πού είναι τα 8 κριτήρια του 2008 και η συμφωνία για την εμπορία των όπλων που έχουν επικυρώσει όλε οι χώρε. Αυτά μπορεί εσά να σα φαίνονται λεπτομέρειε, για μένα έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτά. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντέψκι, για την υπομονή του και για τη δουλειά του. Επανέρχομαι και στην ηθική αυτή τη πρόταση τα ανέφεραν και η Επίτροπο και ο εισηγητή, αλλά πολιτικά θέλω να πω ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία θα το θυμάται αυτό. Από το 54, το 1954 προσπαθούμε και όμως δεν καταφέραμε να έχουμε την κοινότητα άμυνας και τώρα το 2019 επανερχόμαστε και προσπαθούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις αυτής της κοινότητας που απέτυχε. Τώρα λοιπόν όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν εμπιστοσύνη, δείχνουν αλληλεγγύη. Να μην υπάρχει επικάλυψη σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης στην άμυνα, μείωση του κόστους, η οικονομία κλίμακος. Το γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο όλο και περισσότερο αβέβαιο, με μεγάλη αστάθεια, καλό είναι να μπορούμε να διασφαλίζουμε την προστασία μας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Ταμείο αυτό θα μας επιτρέψει καλύτερη ενσωμάτωση των εργαλείων των αμυντικών θα μας βοηθήσει να κάνουμε οικονομίες και θα υπάρξει και μία παρετέρω ολοκλήρωση. Κρίμα που υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες σαν στόχο έχουν να εμποδίσουν τη συμφωνία σε τριμερή διάλογο. Κι όμως είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και μας εκπλήσει που ένα τόσο σημαντικό θέμα τελικά το χειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη σε μια περισσότερο δυνατή Ευρώπη. Ας φροντίσουμε να έχουμε μια πιο δυνατή Ευρώπη που να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους πολίτες της. Να έχουμε αυτό το αμυντικό ταμείο ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την δικιά μας την κυριαρχία, την βιομηχανική και την αμυντική και συγχρόνως να διασφαλίσουμε και την προστασία των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ρικέ. Στη συνέχεια, εκ μέρους της ΓΚΟΕ, έχουμε τη Μαρίσα Ματίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα και μπορείτε να μιλάτε για χρηματοδότηση, αλλά να δώσουμε 13 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα σημαίνει ότι αφαιρούμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα σημαίνει ότι θα ανταλλάξουμε την ελληνική, τη συνοχή, τα μέτρα που προστατεύουν την ποιότητα ζωή των Ευρωπαίων πολιτών για να επενδύσουμε σε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Οι τεχνικέ λύσει ε, δεν αποτελούν παρά ε, ουσιαστικά μια πρόφαση για την πώληση όπλων. Χρειάζονται ασφαλή Ευρωπαίοι, όμως στην απασχόληση, στις δημόσιες υπηρεσίες, σε ένα βιώσιμο μέλλον τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στον τομέα της άμυνας. Με τον ίδιο τρόπο, τίποτα δεν αιτιολογεί να δημιουργηθεί ε, μια νέα γραμμή του προπολογισμού ε, που ούτε καν σέβεται τα όσα εγγράφονται στη συνθήκη είναι μια πολύ ακριβή επιλογή και πολύ πιο ακριβή από τα 13 δισεκατομμύρια που έχουν εγγραφεί εδώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ματίας. Στη συνέχεια για τους πράσινους ο κύριος Μπουτικόφερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός ότι στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την κοινή ασφάλεια. Αυτό είναι το σημείο κίνησης της επιχειρηματολογίας μου. Γι' αυτό λοιπόν ένα αμυντικό ταμείο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίξει ε, θετικό ρόλο. Όμως σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις δεν πετύχαμε το εφικτό. Η επικάλυψη, η ανεπάρκεια θα εξακολουθούν να υπάρχουν στην ε, αγορά των εξοπλισμών το γεγονός ότι σπαταλήσαμε την ευκαιρία που μας προσφέρθηκε. Αυτό ε, δεν οφείλεται στον εισηγητή ε, που θέλω να τον επενέσω γιατί πραγματικά ε, είναι πνεύμα αντιλογίας, πρέπει να το πω αυτό και μερικές φορές μου έκανε και κέφι το να διαπληκτίζουμε μαζί του για το θέμα της πραγματικότητας και του ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων, από τον κύριο Ρουκέ και από την κυρία Γκροστέτ άκουσα ξεκάθαρα του είδα να εκπροσωπούν την, τα γαλλικά λόμπι εξοπλισμών και την ε, στρατιωτικοποίηση, τη σχετική ιδεολογία. Αυτό λοιπόν που έχουμε τώρα είναι ένα αμυντικό ταμείο ε, του οποίου η δεοντολογία και οι αρχές περιοντολογίες είναι απλά μία βιτρίνα. Ένα αμυντικό ταμείο που πολύ σωστά είπε ο κύριος Μαρτά, ε, ένα ταμείο σε 7 χρόνια θα διαθέσει 13 δις. Ένα αμυντικό ταμείο που θα οδηγήσει τελικά ε, στο να έχουμε περισσότερες εξαγωγές εξοπλισμών. Ένας τέτοιος ευνουχισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι όνειδος. Αλλά παρόλα αυτά σημειώθηκε μια καλή ουσιαστική επιτυχία ότι δεν θα δοθούν χρήματα για τους, ε, για τα ρομπότ δολοφόνους. Δεν αρκεί όμως αυτό. Και γι' αυτό εμείς ε, θα καταψηφίσουμε. Κατά τα άλλα, να σας προειδοποιήσω για άλλη μια φορά όσον αφορά την ιδεολογία της ε, στρατηγικής αυτονομίας. Όποιος προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, είναι απλά εθεροβάμων. Ευχαριστώ κύριε Μπουτικόφερ. Στη συνέχεια, ο κύριος Μπουλόκ για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Πρόεδρε, προκειμένου να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή Γιούνκερ θέλει να χρηματοδοτήσει έργα άμυνος που θα κοστίζουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ τεχνολογία για τετρών επικοινωνίες με δορυφόρους, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, εποπτεία στη θάλασσα. Συνεχίζει να εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια ολοκληρωτική ένωση και τελικά προς μια στρατιωτική. Η Κομισιόν προσπαθεί να παρουσιάσει αυτή την εξέλιξη που μια ειρηνευτική διαδικασία, όμως είναι σαφόφωνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποστηρικτές της έχουν έναν στρατό κατά νου. Ο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ε, ενθάρρυνε τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Στρατού πρόσφατα για την υπεράσπιση τη Ευρώπη. Πώ μπορεί κάποιο να δημιουργήσει ένα ομοσπονδιακό στρατιωτικό ε, έργο που θα συμμετέχουν 27 ε, κράτη και 24 γλώσσε, ε, όπω συνήθισε να λέει η Μάργαρετ Θάτσερ, δεν έχει χρήματα παρά τα χρήματα που κερδίζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή που, τη στιγμή που είναι σε κρίση το ευρώ και γίνονται περικοπές για την ανάπτυξη, ε, τώρα, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας τη ε, βιομηχανία ανησυχεί τους πολίτε όπως και διαιρεί άνθρακα. Ένα πανευρωπαϊκός στρατός ε, θα είναι η τελευταία ευρωπαϊκή καταστροφή. Σε αντίθεση με τη Ρωσία ή τη ΗΠΑ, δεν είναι ένας νέο παράγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε και την ψηφοφορία για το Brexit ε, και ε, την ε, κυβέρνηση της Ιταλίας που θα αποθαρρύνουν την περαιτέρω ομοσπονδιοποίηση. Εδώ έχουμε ένα σύνολο γραφειοκρατών που λαμβάνουν αποφάσεις για την άμυνα, για τον πόλεμο και την ειρήνη. Εμεί είμαστε κατά της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού στρατού και ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα συνειδητοποιήσουν ότι να δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Κομισιόν είναι λάθος και είναι η τελευταία μου ομιλία σε αυτό το κοινοβουλίο και ε, απευθύνω έκκληση να απομακρυνθείτε από ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος και δεν θα υπάρξει κανένα καλό από τη Δημιουργία Στρατού και ελπίζω ότι οι εκλογές για το νέο κοινοβούλιο θα ανατρέψουν αυτή την τάση και θα προωθήσουν το σεβασμό του έθνους κράτους και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουλόκ. Και Καλή επιτυχία για το μέλλον. Να σας ευχηθώ. Στη συνέχεια περνάμε στον κύριο Μπούζεκ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον αμυντικό πυλώνα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι η βιομηχανία άμυνας δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά είναι και η ανάπτυξη της βιομηχανίας γενικότερα στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είμαι ικανοποιημένο όχι μόνο λοιπόν για την ανάπτυξη της άμυνας, αλλά και της βιομηχανίας άμυνας. Περί τίνος πρόκειται. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για την συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεύτερον, πρόκειται για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης και πρόκειται και για ενθάρρυνση των χωρών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους σε σχέση με τις παραγγελίες και τις προσφορές. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα στην δικιά μου την περιφέρεια. Έτσι θα μπορέσουμε, πιστεύω, σύντομα να κάνουμε τους Ευρωπαίους να υποφεληθούν από τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα έχουν δημιουργηθεί από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της δικιάς μου περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντεύσκη, ο οποίος πάρα πολύ καλά βοήθησε στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συνεισηγητές, όπως επίσης και την κυρία Γκροστέτ, η οποία ήταν προηγουμένως η συγγήτρια της δικιάς μας έκθεσης για το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πούσεκ, ο επόμενος, ο Βίκτορ Μποστινάρου. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία, κυρία Επίτροπε, να ξεκινήσω από εσά. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τον εξαιρετικό τρόπο που διαπραγματευτήκατε σε έναν κόσμο που έχουμε αστάθεια και πολλέ υβριδικέ και νέε απειλέ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παγιώσει το ρόλο τη ω παγκόσμιο που θα ασκεί επιρροή. Σήμερα η πολιτική Τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την άμενα αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για όλους τους πολίτες μας και γι, αυτή, αυτό βρήκε απήχηση. Η ανάπτυξη της κοινή πολιτικής άμυνας είναι μία από τις κύριες συνεισφορές στην εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκόπος της νομοθετικής πρότασης που έτυχε διαπραγμάτευσης με το Συμβουλίο είναι να ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, έτσι ώστε να απαντήσει στις αυξανόμενες προτεραιότητες της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να να αρχίσουμε να ε, απαντάμε στον κατακαιρματισμό του τομέα της άμυνας ε, και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, ε, να ενθαρρύνουμε την ε, συνεργασία και την κοινή απόκτηση εξοπλισμών. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, είχαμε κύριες προτεραιότητες κλειδί της δικής μου πολιτικής ομάδας για το τομείο αυτό. Εμείς αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αμυντική βιομηχανία και στην πρόθεση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ε, για ε, τα μέσα άμυνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι να υπογραμμίσω την ανάγκη να συνεχίσουμε τη διαδικασία της ε, προώθησης μιας παγκόσμιας τάξης βάσει κανόνων, έτσι όπως αναφέρεται στην Χάρτα 1 και να παγιώσουμε τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, καθώς αυτό αποτελεί τη μόνη εγγύηση ασφάλειας στην Ήπειρό είχα την, ε, ε, το προνόμιο να εργαστώ στο φάκελο αυτό τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να σας συστήσω να υπερψηφίσετε αύριο και καθώς αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο κοινοβόλιο, επιτρέψτε μου να πω σε όλους σας ευχαριστώ καρδίας για αυτά τα 12 χρόνια τα οποία εργαστήκαμε για το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Κυρία Γκροστέτ, ας ε, παραμείνουμε ειρηνικοί αλλά ποτέ αγαθοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 13 δισεκατομμύρια ευρώ τόσα ε, θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ε, μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων σε 7 χρόνια. Αυτά αφαιρούνται από τις επενδύσεις στην καταπολέμηση στόχια, την πρόθεση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Είναι πόροι που θα προωθήσουν τώρα τον πόλεμο, θα χρηματοδοτήσουν την εξοπλιστική βιομηχανία, τροφοδοτώντα μια κούρσα στρατιωτικοποίησης. Ε, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ανοίγεται και την πότρη του προγράμματος έρευνας ε, για, όχι αποκλειστικά για ε, και μη στρατιωτικούς σκοπούς και θα χρησιμοποιήσετε τα δίκτυα μεταφορών για τη στρατιωτική κινητικότητα. Όποιος προωθεί τον πόλεμο και τροφοδοτεί αυτή τη βιομηχανία δεν μπορεί να πετύχει την ειρήνη. Έτσι λοιπόν αυτή η νομοθεσία δεν σέβεται ε, τους λαού. Ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο συνεργασία που να έγκυται στι ε, αξίε της Ειρηνή. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Φεραίρα. Και τώρα ο κύριος Μπουτικόφερ έχει θέσει μια μπλε κάρτα. Δέχεστε παρακαλώ. Κύριε Φερέιρα, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Σας μιλώ φιλανδικά. Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερέιρα, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι στραφήκατε κατά της ε, στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε ότι η δική σας η πολιτική ομάδα, η ΓΚΟΕ, σε όλες αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις των πολλών μηνών δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά ένας έστω ευρωβουλευτής για να συζητήσει. Και ε, δεν καταλαβαίνω πώς τολμάτε να στρέφεστε κατά του μιλιταρισμού και δεν έχετε κάνει τα μαθήματά σας. Κύριε Μπουτικόφερ, αύριο θα επιβεβαιώσετε ότι δεν θα είναι με την υποστήριξη αυτή τη ομάδα που αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα που θέλει να διαθέσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στην εξοπλιστική μηχανία θα εγκριθεί. σω ε, με κάποιε ψήφου από τη δική σα πλευρά, δεν ξέρω, θα δούμε. Σίγουρα με τι ψήφου τη Σοσιαλδημοκρατία και όλη δεξιά. Και φυσικά δεν αγνοώ τη σύνθεση αυτού του οίκου, όπω και εσεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι θέσει μα είναι μη ψηφικέ ακόμη. Και λέω ακόμη γιατί νωρίτερα ή αργότερα και μάλλον νωρίτερα θα είναι πλειοψηφικέ ε, απόψει ε, και εμεί θα ανατρέψουμε αυτή την κούρσα εξοπλισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι εσεί κάπω έχετε ανεχθεί στο παρελθόν αυτέ τι στρατιωτικέ περιπέτειε. Ο κύριος Ταρέν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον ε, συνάδελφό μου, κύριο Μπίτι Κόφα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι παρότι άσκησε κριτική κατά αυτής της πρότασης και σωστά έπραξε, φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι το Ευρωπαϊκό Αμοντικό Ταμείο έρχεται ε, πολύ καθυστερημένα και είναι και πολύ λίγο γιατί δεν κατορθώσαμε να νομοθετήσουμε για να υπάρχει μια, ε, ε, ένας ευρωπαϊκός στρατός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, υποστηρίζω την έκθεση όσον αφορά την αίρεσιμότητα, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Ε, προς τον κύριο Μπούλοκ ε, θα ήθελα να πω ότι η ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Στρατός ε, θα υπάρξει, θα μιλάει αγγλικά. Δυστυχώς ε, λόγω αυτής της περιπέτειας του Brexit δεν θα υπάρξει Βρετανός διοικητής, αλλά θα υπάρξει αυτός ο στρατός. Και προς τον κύριο Φαρέρη, θέλω να πω ότι τα τρία δις είναι τίποτα, ψίχουλα. Ακόμα και ο προπολογισμό ε, της ε, Λετωνίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία αύριο για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο έρχεται στο τέλο μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία. Και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που μα οδήγησαν μέχρι εδώ. Εγώ ήμουν και ο εισηγητή, αλλά θέλω να ζητήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ελέγχει ε, την ε, εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου. Αύριο δεν είναι το τέλο, αλλά είναι η αρχή μια ε, νέα αμυντική πολιτική. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να είναι παίκτη και όχι παρατηρητή. Εγώ είμαστε, ήμουν υπέρ και γενικά η δική μα ομάδα ήταν υπέρ των ε, κατεξοδότηση πράξεων. Ορισμένε τροπολογίε ε, πέρασαν το, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να υψώνει τη φωνή του για να υπάρχει ένα ε, όραμα πραγματικά ευρωπαϊκό που θα επιτρέπει τρία στάδια με πνεύμα του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, τεχνολογίες μας. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να μην υπάρχουν ε, άμεσες απευθείας αναθέσεις. Ε, εμείς έχουμε εκφράσει επιφυλάξει για κάποια κριτήρια, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν χωρίς τιμωρητική διάθεση. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρηματοδοτεί λάθους δεν θέλουμε να υπάρχει συνεργασία με άλλους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά την παραγωγή και την έρευνα. Δεν θέλουμε ε, να διαταράσσεται η αλυσίδα παραγωγής ε, με το να αποκλείονται κάποιες χώρες. Ε, επίσης δεν θέλουμε σε τελική ανάλυση αυτό το ταμείο να ε, χρηματοδοτεί θανατηφόρα όπλα χωρίς ελεγχό η πρόεδρος διακόπτη. Ο κύριος Καστάντο μιλάει με ένα ρυθμό απίστευτα γρήγορο. Πάση περιπτώσει, θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα για έναν ευρωπαϊκό στρατό, ακόμα και εάν ε, ε, αναφέρονται οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου στις συνθήκες. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αυτό το ταμείο, ένα ταμείο το οποίο θα διευκολύνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα διευκολύνει την άμυνα και την ε, ασφάλεια, ένα ταμείο το οποίο δεν θα στρέφεται κατά άλλων, αλλά ούτε θα θέλει να προστατεύει ιδιαίτερα κάποιους, ένα ταμείο το οποίο θα είναι ανοιχτό για άλλες συνέργειες. Τέλος, το ταμείο αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα κενά να ξεχνάμε ότι οι τελικοί χρήστες θα είναι οι δικοί μας οι άνδρες και οι γυναίκες και όλοι εκείνοι που βρίσκονται και σε καθεστώς πολέμου. Πρόεδρος. Ε, κοιτάξτε, οι διερμηνείς πραγματικά τώρα εξεπέρασαν τον εαυτό τους, γιατί δεν υπάρχει και όριο στην ταχύτητα. Μιλάτε τόσο πολύ γρήγορα. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο, ε, πιο αργό ρυθμό, λέει η πρόεδρος επόμενος ομιλητής ο κύριος Γκάλερ. Παρακαλώ κύριε Γκάλερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά έτσι ώστε οι πολίτες μας να προστατεύονται από εξωτερικές απειλές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό το ταμείο ε, για να μπορεί να αξιολογηθεί η ασφάλεια και να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το βρίσκω πάρα πολύ λυπηρό το ότι κάποιοι από αριστερά αλλά και μέχρι δεξιά ε, δεν θέλουν να προσφέρουν αυτή την καλύτερη προστασία στους πολίτες μας. Αυτό είναι ολιγορία. Ολιγορία κατά των πολιτών στρατιωτών μας που τους αξίζει καλύτερη άμυνα ολιγορία και έναντι των στρατιωτών μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή παρήματος χάρη στο Μαλί, ε, στη Σομαλία, στη Μεσόγειο υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας. Έχουν το δικαίωμα να έχουν τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίζουν υγιείς στις πατρίδες τους. Τέλος, αναφέρομαι στο Συμβούλιο και στα μεμονωμένα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή. Στο μέλλον εσείς θα κληθείτε να αποδείξετε δείξετε ότι τα 13 δι που προβλέπονται για τον αμυντικό αυτό προπολογισμό θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού για αγορές, ε, για εξοπλισμούς, ε, για βελτίωση τη ικανότητας. Τώρα πρέπει να αποδείξετε ότι ε, τα 210 δι ευρώ στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται καλύτερα οι πρωτεύουσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και όχι να θέλουν να καταφύγουν σε προγράμματα όπως το ΕΦΚΑΣ ή τα τεθωρακισμένα μάχης. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες μας τελικά τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Από το σύνθημα στρατηγική αυτονομία θα πρέπει να περάσετε σε μια συνεπή αμυντική πολιτική, πολιτική εξοπλισμών έτσι ώστε οι πολίτες μας και η βιομηχανία μας να κατανοήσουν κατανοούν περί τίνος πρόκειται. Ε, το ταμείο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι το, μόνο το πρώτο βήμα και κατά τα άλλα θα χαιρόμουν πάρα πολύ ε, το πώς θα, να δω πώς θα ψηφίσω ο κύριος Μπούλμαν από τον ε, πρόεδρο μια τόσο μεγάλης πολιτικής ομάδας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Μπορεί κανείς να περιμένει και μια προσωπική τοποθέτηση. Ο κύριος Ροζάτης στη συνέχεια για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα συζητάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ασφάλεια της Ευρώπης, ε, μια αγορά δημόσιων κονδυλίων ε, για την απόκτηση αμυντικών μέσων. Αυτό είναι κατακαιρματισμένο ε, στην Ευρώπη. Μόλις το 16% αυτών των ε, δημόσιων διαγωνισμών υλοποιούνται από δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επίπεδο συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο. και φυσικά ε, η ασφάλεια αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας και υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις ε, όπως η επιθετική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ο μουσουλμανικός ε, εξτρεμισμός και απαιτούν να ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ακριβώς αποτελεί ένα μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία στο βιομηχανικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη του κλάδου στα κράτη-μέλη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει 13 δισεκατομμυρία ευρώ. Ένα ποσό που θα επιτρέψει την ενίσχυση των ικανοτήτων ε, στην έρευνα και στην κοινοτομία, στον αμυντικό κλάδο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην κατανομή των κορδιλίων ε, για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε το δυναμικό όλων των χωρών και αναφέρομαι και στις μεγάλες χώρες αλλά και στη χώρα μου, στην Πολωνία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωσάτη. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Κατσδιάη. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Πόσπεσιλ πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσωπικά όλη τη συζήτηση και θα την στηρίξω. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Αυτές οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό γενικότερα για την οικονομία. Τέτοια προγράμματα δεν είναι δυνατόν βέβαια να απειλούν τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να αποτελούν μια εναλλακτική λύση διαφορετική από το ΝΑΤΟ. Εμείς στην Τσεχία πιστεύουμε ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασίας. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση, αλλά η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ να ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Πρώτος, ευχαριστούμε κύριε Πόσπισιλ. Ο κύριος Μαριάς τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 13 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αντιμετώπιση της φτώχειας. θεωρώ ότι αυτό το ποσό επί της ουσίας θα μπει στην υπηρεσία των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών της ευρωπαϊκής ένωσης που ως γνωστόν πουλάνε όπλα ακόμη και στην τουρκία ακόμη και στη σαουδική αραβία. στην πράξη τι γίνεται; ζήτησε ο τραμπ να βάλει η ευρωπαϊκή ένωση το χέρι στην τσέπη για τα θέματα της άμυνας. αυτό είναι όλο το θέμα. και πλέον ερχόμαστε να υπηρετήσουμε αυτή την πολιτική μετατρέποντας σε όλο και πιο στρατιωτικοποιημένη την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση και γι' αυτό αυτό που θα συμβεί στην πράξη είναι να γίνονται όλο και πιο πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης στον τρίτο κόσμο. θεωρώ ότι τα κονδύλια αυτά πρέπει να πάνε κυρίως για τη στήριξη της ίδιας της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Παρακαλώ. Κύριε Σόσνιερτς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε αυτά που είπε ο καθηγητής Κρασνοντεύσκη, ότι πρόκειται για ένα παραπάνω βήμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας. Και αρκεί να ακούσουμε την κυρία Κροστέτ για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία σε βάθος ολοκλήρωση. Καταλαβαίνω ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να πετύχουν περισσότερα. Χάσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε τώρα βρίσκονται στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και δρούν ανάλογα. Πώς όμως θα υποφεληθεί η Πολωνία. Ουσιαστικά καταστρέφουμε την ανεξαρτησία μας. Χάνουμε τον έλεγχο του δικού μας ε, στρατού. Η έρευνα και ανάπτυξη που μπαίνουν ε, σε κοινό πλαίσιο σημαίνει ότι χάνουμε τον έλεγχο της δικιάς μας έρευνας και ανάπτυξης. Τι θα γίνει στις χώρες οι οποίες τελικά δεν θα έχουν το δικό τους στρατό. Φτιάχνουμε ένα τέταρτο ράιχ της Γερμανίας. Πρόεδρος, τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, με ευρωβουλευτές, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τίποτα δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή, δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους που με τόση αφοσίωση προσπαθήσετε να ε, καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Σε δύο πτυχές θα αναφερθώ μόνο. Πρώτον, για τη συνεργασία, γιατί πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο ποσό, στα χρήματα. Θέλω να σας πω και πάλι ότι η έλλειψη συνεργασίας στον τομέα της άμυνας κοστίζει και το κόστος αυτό είναι ανάμεσα στα 25 με τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, επειδή δεν υπάρχει συνεργασία στον αμυντικό βιομηχανικό τομέα. Έπειτα, για την εξαγωγή όπλων, επειδή κάποιοι από εσά το έθεσαν. Και εδώ είναι σαφές το θέμα. Έχουμε συζητήσει πολύ γι' αυτό. Είναι καθαρά αρμοδιότητα των χωρών μελών. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα με τον κανονισμό. Δεν αυξάνουμε την εξαγωγή όπλων. Αυτό που θέλουμε και αυτή που είναι η πρόθεσή μας είναι να μειωθεί η εξάρτησή μας από